Επίσης δεν βλέπω να υπάρχουν και έτσι η εντολή αυτή επικυρώνεται. Η υπογραφή πράξεων νομοθετικού χαρακτήρα που αφορούν την κανονική διαδικασία που κινούμε τον πρόεδρο του Συμβουλίου την Τετάρτη θα υπογράψω πέντε νομοθετικές πράξεις όσον αφορά το άρθρο 74 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δημοσιευθούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης αυτές οι προτάσεις. Από το ΕΛΚΑ και την Προοδευτική Συμμαχία Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβα τους ε, διορισμούς ε, σε